τις υπηρεσίες, έλλειψη προόδου στο Συμβούλιο και καθυστέρηση της Επιτροπής όσον αφορά την έγκριση ορισμένων προτάσεων. Να σας πληροφορήσω πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση ότι για τη συζήτηση αυτή δεν προβλέπεται η διαδικασία της μπλε κάρτας. Λοιπόν, δίνω αμέσως το λόγο στην κυρία Μπόλς για ένα πεντάλεπτο. Ευχαριστώ. Κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας είχαμε κατακλυσμό νομοθετημάτων για τις μοτοτικές υπηρεσίες. Από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την το FMD, ξεκινήσαμε και τη δημιουργία τη Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή και περάσαμε από διάφορα μέτρα για την αγορά και τι τράπεζε, προστασία επενδυτών και καταθετών και με, με αναμένεται ακόμα μηχανισμό επιλύσεω των προβλημάτων. Πάνω από 40 πρωτοβουλίε έχουν ολοκληρωθεί ή έχουν δρομολογηθεί ή αναμένονται σύντομα. Η Επιτροπή ΕΚΟΝ επί μακρόν ζήτησε αξιολόγηση συνεπιών όσον αφορά τη νομοθεσία για τα χρηματοστατικά και παρόλο που έχουν ολοκληρωθεί πολλά, υπενθυμίζω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι έχει υποχρέωση να κάνει ανάλυση κόστο ωφέλου όσον αφορά την αλλαγικότητα και την αποτελεσματικότητα τη υιοθετηθή νομοθεσία από την αρχή της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Αυτό είναι κάτι που ξεκινήσει τώρα και να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος αυτής της θητείας. Θα γνωρίζετε ίσως, Επίτροπε, ότι η Επιτροπή ΕΚΟΝ ξεκίνησε τη δική της δεύτερη έρευνα και συλλέγει στοιχεία τώρα. Τώρα όσον αφορά τον ροή των εργασιών, δύο πράγματα ήταν χαρακτηριστικά. Καταρχάς, πολλές προτάσεις ε, οδήγησαν σε μεγάλη καθυστέρηση χρονική από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν κάποιε δικαιολογίε, αλλά παραμένει γεγονό ότι υπήρξαν μακρέ καθυστερήσει, όπω για το μηχανισμό επιλύσεω των προβλημάτων και εξυγίανση, κάτι που ήθελε το Κοινοβουλίο, όπω και το ίση το 2009 και την οδηγία για την ομοθεσία για τα αξιόγραφα. Αυτά τα θέματα έχουν δύσκολα προβλήματα νομικής φύσεως και γι' αυτό το λόγο ε, πρέπει μάλιστα να υποβάλλονται έγκαιρα ώστε οι συνομοθέτες να μπορούν να εργαστούν. Ε, δεύτερο χαρακτηριστικό των εργασιών ήταν ότι το Κοινοβούλιο εργάστηκε γρήγορα ε, και πυρετοδό, δίνοντα πληροφορίε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν προτείνει νομοθετήματα και ε, σε αντίδραση διαβουλεύσεων κινήθηκε πάρα πολύ πιο γρήγορα από το Συμβούλιο. Λοιπόν, τώρα έχει, υπάρχουμε χρονική καθυστέρηση, περιμένουν σημαντικέ προτάσει και οι προτάσει αυτέ έχουν πολύ λίγε πιθανότητε να συζητηθούν στον τριμερή διάλογο. Για άλλα νομοθετήματα, λόγω λήψεω συνένεση στο Συμβούλιο, το Συμβούλιο χρονοτριβεί παραδείγματο χάρη για το MIFID και τις ε, κεντρικά σημεία καταθέσεων αξιογράφων. Ε, και φαίνεται τελικά ότι είναι, πρέπει να πολεμήσουμε διάφορα τέρατα στο Συμβούλιο και εδώ. Λοιπόν, πρέπει να προχωρήσει το Συμβούλιο τόσο ώστε να ξεκινήσουν οι τριμερείς διάλογοι και προειδοποιώ, κοιτάξτε τις θέσεις του Κοινοβουλίου, διότι δεν θα υποχωρήσουμε ε, στην γραμμή που ακολουθεί το Συμβούλιο που λέει ότι πρέπει να επιτευχθεί ευαίσθητη ισορροπία στο Συμβούλιο. Όσο απογοητευόμεθα από την κολυσιεργία και ότι κολλάνε προτάσει στο Συμβούλιο, τόσο θα είμαστε αποφασισμένοι εμεί να επιμένουμε στι θέσει μα ε, στα θέματα αυτά που φτάνουν στον τριμερή διάλογο. Στη συνεδρία συντονιστών χτε στην ΕΚΟΝ ε, συμφωνήθηκε ότι δεν θα χαλαρωθεί η θέση μα παρά τι επικείμενε εκλογέ. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμεθα επί όλων των θεμάτων όσων αυτά καταφθάνουν Πέραν ολοκληρώνοντας τις πρώτες αναγνώσεις επί όλων των προτάσεων που είναι επιτάπητο σε αυτή τη φάση. Ε, κατανοώ ότι χρειάζεται θέσεις προτεραιοτήτων και ότι το να κάνει κανείς λίγο από τα πάντα και να ολοκληρώνει τίποτα δεν είναι αυτό που πρέπει να γίνεται ε, τώρα προς το τέλος της θητείας. Όμως περιμένουμε να διπλασιαστούν οι προσπάθειες του Συμβουλίου για τις ε, εκκρεμούσες προτάσεις ώστε οι περισσότερες από αυτές να τύχουν συμφωνίας πριν από το τέλος της θητείας αυτού του Κοινοβουλίου. Η Τραπεζική Ένωση βεβαίω αποτελεί προτεραιότητα για τη σταθερότητα και των τραπεζών και των ε, κρατικών ομολόγων και γι' αυτό θέλουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θετήσει γρήγορα προτάσει τη, ώστε να υπάρξει ένας ενιαίος μηχανισμός για επίλυση αυτών των προβλημάτων και πρέπει να ολοκληρωθεί και εργασία όσον αφορά τι κεφαλικέ απαιτήσει για τι τράπεζε και την επίλυση προβλημάτων των τραπεζών και ζητούμε να ακολουθηθούν οι συστάσει τη ομάδα Λικάνεν όσον αφορά τι δομικέ μεταρρυθμίσει των τραπεζών. Και ξεχνά, ξαναλέω ότι υπάρχει έλλειψη κρίσεων όσον αφορά την οδηγία για ταξιόγραφα. αξιόγραφα. Ήδη, όπω είπε επανειλημμένα, απευθυνόμενοι προ την λουθενική Προεδρία που επίκειται. Η πρόσβαση στου τραπεζικούς λογαριασμούς είναι ύψιστη προτεραιότητα για πολλούς πολίτες. Ξοδέψαμε χιλιάδες ωρών για θέματα οι μεγάλε επιχειρήσει και μεγάλους χρηματοδοτικού φορείς. Τώρα πρέπει να δείξουμε ότι θα προσέξουμε όλους όλα τα μέλη της κοινωνία, δίνοντα πρόσβαση σε αυτό το ζωτικό εργαλείο τη σύγχρονη ζωή, τον τραπεζικό λογαριασμό. Θα ήταν το για το Συμβούλιο αυτό να τα αφήσει παράμερα, θεωρώντα το λιγότερο σημαντικό. Πρέπει να γίνει αυτό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για το Συμβούλιο. Υπουργό, ε, κυρία Κρέιτον έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε αξιότιμα μέλη με ιδιαίτερα ευγνώμων για την ευκαιρία να λάβω μέρος σε αυτή τη συζήτηση σήμερα και να διευκρινίσω ορισμένα σημεία. Ελπίζω ότι αυτό θα επιτρέψει σε όλους να προχωρήσουμε και να βελτιώσουμε τη συνεργασία μας σε αυτό τον τομέα. Πρώτον, δεν μπορώ να συμφωνήσω με το θέμα πάνω στο οποίο βασίζεται η ερώτηση. Υπάρχει έλλειψη προόδου ό,τι αφορά τον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών το Συμβούλιο εξακολουθεί να σημειώνει σημαντικές προόδους στα πλαίσια δύσκολων διαπραγματεύσεων για το θέμα αυτό. Μέχρι στιγμής έχουμε δώσει προτεραιότητες στο θέμα του τραπεζικού τομέα, κάτι που δικαιολογείται λόγω της σημασίας αυτού του τομέα και της ανάγκης να προωθηθούν αυτά τα θέματα. Έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδο στον τομέα των χρηματοπιστωτικών θεμάτων. Έχουμε καταλήξει σε μια συμφωνία για τη μεταρρύθμιση του τραπεζικού τομέα και για τη μελλοντική τραπεζική ένωση. Το θέμα της εποπτείας των τραπεζών και το θέμα των κεφαλαϊκών απαιτήσεων οι σχετικοί κανονισμοί και έχω αναφερθεί στη σημασία αυτών των νομοθετικών κειμένων κατά επανάληψη και αποτελούν σημαντικές προτεραιότητες από την αρχή του, της Προεδρίας μας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αναβάλει μέχρι το Σεπτέμβριο την ε, ψηφοφορία και ελπίζω ότι αυτή η αλλαγή δεν θα εμποδίσει την ολοκλήρωση των εργασιών. Έως ότου εγκριθεί από τα δύο ε, ε, σώματα, για να γίνει αυτό οι διαπραγματεύσει θα δύσκολες. Τελικά καταλήξαμε σε μια συμφωνία για το θέμα των των στεγαστικών δανείων και ελπίζω ότι αυτή η οδηγία θα εγκριθεί μετά την πρώτη ανάγνωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εφόσον θα τηρηθούν οι συμφωνίες του 2011 πρόσφατα καταλήξαμε σε πολιτική συμφωνία σε ό,τι αφορά την οδηγία για τη διαφάνεια που θα κάνει πιο ελκυστική, πιο ελκυστική την αγορά ε, ε, για τους μικροκαταθέτες την, την τραπεζική αγορά. Υπάρχουν και άλλα θέματα επιτάπητος, αλλά πρέπει να μιλήσουμε για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Έχουμε περίπου 20 νομοθετικές προτάσεις για τον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και καθώς, καθώς θα καταλήγουμε σε συμφωνία με ορισμένες θα συνεχίζονται οι προσπάθειες δεν υπάρχει λόγος να διατυπώνουμε νέες προτάσεις, λέει ο Επίτροπος Μπαρνιέ. Σωστά, αλλά οι προτάσεις της Επιτροπής και οι μελαγές που προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χρειάζονται περαιτέρω επεξεργασία. Απαιτείται συζήτηση, διαβούλευση και πρέπει κατόπιν να εγκριθούν. Γι' αυτό πρέπει να ε, αξιοποιήσουμε την εμπειρία που υπάρχει στα κράτη-μέλη. Θέλουμε να προσφέρουμε νομοθεσία υψηλού επίπεδου που θα είναι αποτελεσματική και εφαρμόσιμη. Θέλουμε να προχωρήσουμε γρήγορα χωρίς να θυσιάσουμε την ποιότητα στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας. <clears throat> Ένα παράδειγμα είναι η διαδικασία αναθεώρησης του ΜΥΦΙΔ που αποτελεί τον ακρογωνιαίο ε, λίθο για την ολοκλήρωση της ε, τραπεζικής αγοράς. Πρέπει να προωθηθούν τεχνολογικές εξελίξεις, οικονομικές ε, καινοτομίες και όλα αυτά πρέπει να εφαρμοστούν με αποτελεσματικό και σωστό τρόπο για να καταλήξουμε σε ένα πιο ισορροπημένο, ισορροπημένο κείμενο που είναι κάτι που δεν μπορεί να δημιουργηθεί μέσα σε μία νύχτα και επίση και το θέμα των εγγύσεων. Η προσέγγιση που έχουμε επιλάξει είναι να ολοκληρωθούν οι ρυθμίσει για την εξυγίανση των τραπεζών σε ό,τι αφορά, στο και να λάβουμε επίση υπόψη και το θέμα της προστασίας των καταθέσεων. Ε, ε, είναι λογικό να, να αφήσουμε κατά μέρος προς το παρόν την πρόταση DGS. Το ίδιο το Κοινοβούλιο επέλεξε να ψηφίσει για το θέμα αυτό το 2012 και το Συμβούλιο συνεχίζει συστηματικά τις προσπάθειές του στα πλαίσια του τριμερούς διαλόγου. Οι διαπραγματεύσεις αυτές θα χρειαστεί να περιμένουν έως ότου υπάρξει για αυτό το θέμα συμφωνία. Έχουμε επίσης αναγνωρίσει τη σημασία να υπάρχει εποπτεία, εποπτεία, εποπτικός έλεγχος αλλά δεν θα μπορέσουμε να συμβάλλουμε άμεσα σε αυτό διότι περιμένουμε πρώτα απ' όλα να γίνει μια αξιολόγηση των επιπτώσεων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η πρόοδος ε, υπήρξε εντυπωσιακή πρέπει να πω. Βεβαίως πάντα υπάρχει περιθώριο για βελτίωση. Το Συμβούλιο θα διατηρήσει το ρυθμό της προόδου και ελπίζουμε ότι θα εξακολουθεί να κάνει το ίδιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. <clears throat> Για το μέλλον ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε για μια ενιαία προσέγγιση σε ό,τι αφορά την οδηγία για την εξυγίανση των τραπεζών και το θέμα των ε, τραπεζικών λιανικών προϊόντων. Θα, θα γίνει μια πρόταση για ένα ενιαίο ε, ε, σύστημα εξυγίανσης μέχρι το τέλος του χρόνου. Θα τηρήσουμε αυτό το χρονοδιάγραμμα στο πλαίσιο και των άλλων προτεραιοτήτων μας. Είχαμε ελπίσει να υπάρξει πολιτική συμφωνία για τον νησμό, αλλά δεν είμαστε τώρα βέβαιοι κατά πόσο οι, κατά πόσο προοπτικές, ποιες θα είναι οι προοπτικές μετά τον τριμερή διάλογο που θα γίνει σε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουμε σημειώσει επίσης προοδούς για το θέμα του αποθετηρίου <clears throat> τίτλων και θα μελετάμε και άλλους φακέλους όπως το UCITS και την πρόταση της Επιτροπής για την, για την καταπολέμηση του ξεπλήματος του βρώμικου χρήματος. Όλοι αυτοί οι στόχοι είναι επιτεύξιμοι. Θα απαιτήσουν την υποστήριξη της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να μπορέσουμε να φτάσουμε τελικά σε έναν αποδεκτό συμβιβασμό. Ολοκληρώνοντας θέλω να πω ότι δεν δέχομαι ότι έχει υπάρξει έλλειψη προόδου από πλευρά Συμβουλίου όπως είπαμε, έχουν σημειωθεί σημαντικές πρόοδοι για πάρα πολλά θέματα, για πάρα πολλούς φακέλους και μιλάμε για θέματα λεπτομερή και σύνθετα. Επιδιώκουμε γρήγορα αποτελέσματα, αλλά θέλουμε και ποιοτικά αποτελέσματα και αυτό πολύ συχνά απαιτεί χρόνο. Ελπίζουμε θα συμβάλλει και θα παίξει το ρόλο του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και προσβλέπουμε σε συνεχές επαφές για τους επόμενους μήνες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο Επίτροπος ο κύριος Μπαρνιέ τώρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους σας. Καταρχάς ευχαριστώ την Sharon Bowles και την Επιτροπή Οικονομικών Ξενοτικών Υποθέσεων για το ερώτημα αυτό. Πιστεύω ότι πρέπει να πω κυρία Πρόεδρε ότι τρία χρόνια και κάτι παραπάνω μετά την αρχή της θητείας, πέντε χρόνια μετά την αρχή της χρηματοστητικής ε, κρίσεως, της φοβερής που ήρθε από τις ΗΠΑ και διαδόθηκε στην Ευρώπη και οι συνέπειες της οποίας ε, πόρα απέχουν από τον τερματιστούν, ήρθε η στιγμή, είναι και η ώρα, το έτος αυτό, το 2013, να δούμε κατά πόσο κάναμε αυτά που είπαμε, τα πραγματοποίησαμε, να αξιολογήσουμε τι καπραγματοποιήθηκε, τι κάναμε και να πούμε με πνευματική διάβγεια πώς πρέπει να προχωρήσουμε από εδώ και πέρα, κυρίως για να λάβουμε υπόψη την οικονομική και κοινωνική κατάσταση ε, και να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν το κοινοβούλιο σας που μου δίνει αυτή την ευκαιρία μέσω της ερωτήσεως να ε, αναφερθώ σε αυτό το θέμα, να κάνω μια αποτίμηση. Το κάνω και έναντι της Λουσίνα Κράιτον και τη Ιρλανδική Προεδρία και ευχαριστώ προσωπικά την Ιρλανδική Προεδρία εκ μέρου και τη ομάδα μου και την ομάδα του Υπουργού Μάικλ Νούναν διότι με αποφασιστικότητα και επιδεξιότητα εργάζονται. Ε, ξεκινήσαμε λοιπόν μαζί κυρίες και κύριοι βουλευτές εδώ και τρία χρόνια, επί εδώ και τρία χρόνια βρίσκομαι σε αυτή τη θέση, ξεκινήσαμε ένα χρονοδιάγραμμα. Η Σάλλον Μπρόλ αναφέρθηκε σε κατακλυσμό νομοθετημάτων. Δεν ξέρω αν είναι σωστή αυτή η παρουσίαση. Ένα πρόγραμμα όμως θα έλεγα πρωτοφανές ε, όσον αφορά τα θέματα χρημα, ρύθμιση, ρύθμισης. Έχω το State of Play, αυτό το μικρό έγγραφο που ξέρετε, ε, τι ψηφίστηκε, τι έχει δρομολογηθεί προς ψήφιση, τι έχουμε μπροστά μας και συζητούμε όσον αφορά τα νομοθετήματα. Γιατί κινηθήκαμε τούτο τρόπος, διότι αυτή η χρηματοπιστωτική κρίση έχει λόγους, έχει αίτια. Και βασικό αίτιο, κατά την άποψή μας, είναι η έλλειψη ρύθμισης σε παγκόσμιο επίπεδο, έλλειψη σωστής εποπτείας. Των τραπεζών επιτρέψαμε στους τραπεζίτες να κάνουν τα πάντα και επέτρεψαν σε αυτούς τους να κάνουν τα πάντα. Με μπόνους πρωτοφανή, ενθαρρύνοντας την ανάληψη κινδύνων, ώστε τελικά να πληρώνει το κίνδυνο ο φορολογούμενος. Ε, έλλειψη κεφαλαίων για τις τράπεζες, δεν υπήρχε εξασφάλιση ρευστότητας. Ε, έπαιξαν ρόλο όλα αυτά. Λοιπόν, όπως ζητήθηκε από τους G20 και όπως χρειάζεται σε παγκόσμιο επίπεδο και ευρωπαϊκό επίπεδο, ο κάθε φορέας από εμά, για κάθε προϊόν, για κάθε τομέα, προσπαθούμε να βρούμε λύση. Κανείς δεν θα ξεφύγει. Κανείς δεν πρέπει να ξεφύγει από ρύθμιση, δημόσια ρύθμιση και ευφυή εποπτεία. Αυτό είναι το πνεύμα τη προσπάθεια που καταβάλουμε και των εργασιών. Και σήμερα, κυρίε και κύριοι βουλευτέ, για κούραση δεν υπάρχει χώρο. Για πάυση, για ανάπαυση. Κάτι που ακούω καμιά φορά. Υπάρχει χώρο, και αυτό είναι το πνεύμα τη προφορική ερωτήσεω τη κυρία Μπόλ, υπάρχει χώρο για επαγρύπνηση, για αποφασιστικότητα και για πραγματισμό, πραγματιστική προσέγγιση όσον αφορά τα κείμενα που υποβάλλουμε. Να αναφέρω για το επόμενο εξάμεινο ποιε θα είναι οι προτεραιότητε πέραν από αυτά που έγιναν. Λοιπόν, η Τραπεζική Ένωση καταρχά. Η Λουσίντα Κράιτον αναφέρθηκε στο θέμα. Θέλουμε πολύ γρήγορα να ολοκληρωθεί το θέμα αυτό βάσει τη προτάσεω που υπέβαλα εδώ και ένα χρόνο, πάνω από ένα χρόνο, για την εξυγίανση των τραπεζών. Και ευχαριστώ τον Γκούναρ Ότμαρ και την Επιτροπή ΕΚΟΝ ε, για την ψηφοφορία που έγινε τον πεσμένο μήνα. Εργαζόμαστε άοκνα, ούτω ώστε στο επόμενο Συμβούλιο Κοφίν 21 Ιουνίου το Συμβούλιο είναι σε θέση να καταλήξει κοινή θέση. Και μετά εμείς βεβαίω να μπορέσουμε να κάνουμε από κοινού την προσπάθεια μαζί με το Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να πω ότι επί τη ευκαιρία του τελευταίου κομματιού, αν θέλετε, του πακέτου για την εξυγίανση, συνεργάζομαι με την ομάδα μου για να παρουσιάσω πολύ σύντομα τι επόμενε εβδομάδε τις επόμενες ημέρες μάλιστα πρόταση που αφορά τον σχετικό μηχανισμό για την εξυγίανση, τον ενίο μηχανισμό που θα χρησιμοποιείται στην Ευρώπη. Θα παρουσιάσουμε αυτή την πρόταση και θα αποτελέσει αντικείμενο επεξεργασίας μαζί με την ε, Λιθωνική Προεδρία. Στο ίδιο πνεύμα μπορούμε πολύ γρήγορα να κινηθούμε σε κάτι που ανέφερα χτες. Το συζήτησα με τον Πίτερ Σάιμον. Το κείμενο για τις ε, εγγύσει για καταθέσεις διότι είναι αλληλένδετα όλα αυτά για την δυνατότητα να υπάρχει πρόληψη των προβλημάτων και να προστατεύονται οι καταθέτες. Δεύτερο εργοτάξιο, ούτως υπήν, μιλάμε για διορθωτικά μέτρα και νομοθεσία, για προληπτικά μέτρα και καμιά φορά μέτρα καταστολής λαμβάνονται, όπως η οδηγία για την κατάχρηση των αγορών Υπουργό αναφέρθηκε προηγουμένω για το κείμενο που έχω στην καρδιά μου, για την καταπολέμηση κατά του ξεπλήματο του χρήματο και των προϊόντων του εγκλήματο. Όλα αυτοί οι νόμοι ανήκουν στην απαιτούμενη αντίδραση και στην υποχρεωτική πρόληψη που πρέπει να επιβάλλεται για να αντιμετωπίζεται η χρηματοστική κρίση. Θα πρέπει να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα αυτό της διορθωτικής ρύθμισης και επιγραμματικά παραθέτω τα όσα έκανε για το μύφιντο Μάρκους Φέρμπερ τη συζήτηση που συνεχίζεται στο Συμβούλιο με μια συμφωνία που επίκειται επί Ιρλανδικής Προεδρίας, ελπίζω, ε, και θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε το διάλογο, τον τριμερή διάλογο επί Λιθουανικής ε, Προεδρίας. Κατάχρηση των αγορών. Αλλά μακάρτι δεν είμαστε μακριά από μια συμφωνία που θα πρέπει να επισημοποιηθεί παράλληλα με το ΜΥΦΙΤ Ανέφερα και με τις συζητήσεις για το Omnibus που θα πρέπει να ξεκινήσουν εκ νέου πολύ σύντομα βάσει συμπληρωματικής μελέτης που ζήτησα από την ΑΙΟΠΑ μια, την Ευρωπαϊκή Αρχή ε, εποπτείας των τραπεζικών, ε, των ασφαλιστικών ταμείων και των συνταξιδικών ταμείων. Τρίτο εργοτάξιο. Πρέπει να περάσουμε από την αντίδραση και την πρόληψη και να καταλήξουμε σε άλλη μορφή ρύθμισης Δηλαδή, πιο ενεργητική, πιο δραστήρια, πιο δυναμική νομοθεσία πρέπει να θεσπίσουμε για να ενθαρρύνουμε και να διευκολύνουμε την ανάκαμψη και την ανάπτυξη μέσω των μέτρων που λαμβάνονται από όλε τι χώρε και σε συλλογικό επίπεδο. Αυτό είναι και το πνεύμα πολλών προτάσεων που έκανα σε αυτό το χρονοδιάγραμμα στο πρόγραμμά μα. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την ε, Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, το Διαβατήριο για τα Κεφάλαια Κινδύνου, προβληματισμό που κάνουμε για την υποστήριξη, την πλαισίωση, την ευφύ πλαισίωση του ε, cloud funding, ε, του συμμετοχή και η χρηματοδότηση. Ε, το κείμενο το ξέρει πως Κρούτε όσον αφορά την διαφάνεια, την τραπεζική συμφωνία, τη διαφάνεια και την τραπεζική κινητικότητα και τη διαφάνεια των τελών που εισπράττουν οι τράπεζες. Και κάτι άλλο που με απασχολεί πολύ, η πράσινη βίβλος που αφορά την μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. Λοιπόν, κρινόμεθα όσον αφορά τη μεθόδο εργασία μας, ε, κυρίες και κύριοι, πέραν τη ουσία, όσον αφορά αυτό το θέμα, είμαστε πιστοί στι απαιτήσει που επεβάλαμε στους εαυτούς μα να μην ε, αυτοσχεδιάζουμε, να εργαζόμεθα όμω γρήγορα, σοβαρά και να θεσπίσουμε νομοθεσία ευφυώ. Πριν από κάθε πρόταση ξεκινάμε συζητήσει και διαβούλευση. Δίνω μεγάλη σημασία σε αυτές τις μελέτες ε, συνεπιών και κυρία Μπόλ, είναι και η ώρα μελέτη ε, σφαιρική, θα έλεγα, ακόμα και αν είχα την ιδέα να την πραγματοποιήσω, δεν μπορώ να την κάνουμε σοβαρά πριν να έχουμε κείμενα τα οποία είναι αρκετά διάφορα στο τέλος νομοθετική διαδικασίας βελτιωμένα σε σχέση με τα αρχικά κείμενα που υπέβαλα κατόπιν συνεργασία μαζί σας. Με βάση λοιπόν κείμενα τα οποία έχουν σχεδόν όλα οριμάσει, ξέρουμε ποια είναι η πραγματικότητα και η ακρίβεια των κειμένων, ήρθε η ώρα να κάνουμε μια σφαιρική μελέτη αντιχτύπου και προσπαθώ να βρω πώ μπορούμε να κινηθούμε γρήγορα και αντικειμενικά για να πραγματοποιηθεί αυτή η μελέτη αντικτύπου, γνωρίζοντα τη σημασία που έχει αξιολόγηση των κειμένων για τη ρύθμιση και για την, για την εξοικονόμηση πόρων γενικά και την οικονομία. Επανειλημμένα είπα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βελτίωσε τα κείμενα αυτά ε, και πέτρεψε την παγίωσή τους. Θα ήθελα να πω κάποια τελικά πράγματα πολύ γρήγορα για τα δύο σημεία που αναφέρατε συγκεκριμένα κυρία Πρόεδρε η νομοθεσία όσον αφορά τα δικαιώματα για τα, για τα αξιόγραφα, το νομοθεσία για τα αξιόγραφα μάλλον, πολύ σημαντικό στα πλαίσια των πολιτικών δικαιωμάτων και τη εθνική νομοθεσία για την ιδιοκτησία. Υπάρχουν μεγάλε αποκλήσει μεταξύ των 27-28 κρατών μελών. Γι' αυτό λοιπόν εξετάσαμε όλους τους εθνικούς κανόνες όσον αφορά ε, αυτά τα θέματα των αξιογράφων. Ε, ήταν μια υποχρέωση αυτή να κάνουμε μια μελέτη πριν θεσπίσουμε, ετοιμάσουμε ένα κείμενο. Ετοιμάζουμε δημόσια διαβούλευση σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τι νομικέ πτυχέ, όσον αφορά ε, το δίκαιο αυτό των αξιογράφων το 2011. Συμμετείχαμε σε διεθνεί ομάδε εργασία που συζήτησαν το θυμιστικό πλαίσιο για τα δάνεια και την ε, χρήση των αξιογράφων απλευρά συνταξιωτικών ταμείων. Ε, συνεχίζονται οι εργασίε όσον αφορά τη μελέτη αντικτύπου ε, πριν να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει νομοθετική πρόταση και ελπίζω αυτό να μπορέσει να γίνει όσον αυτό το θέμα αυτό, κυρία Πρόεδρε, το επόμενο φθινόπωρο. Δεύτερο σημείο, η οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών με ταχικά PLD τις αγορές ε, πληρωμών του λιανικού εμπορίου, του λιανικού τομέα. Ε, υπήρξαν πολλές βελτιώσεις τα τελευταία χρόνια, κυρίως στα πλαίσια των πληρωμών μέσω κινητών τηλεφώνων, καρτών και διαδικτύου. Συνέχεια έχουμε εξελίξεις, δεν ολοκληρώθηκαν προσπάθειες. Από το 2007 χρονολογείται η οδηγία και δεν αντιστοιχεί πλέον στις παρούσες συνθήκες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2012 προέβησε δημόσια διαβούλευση με μια πράσινη όσον αφορά τι πληρωμέ μέσω κάρτα, μέσω διαδικτύου και μέσω κινητού τηλεφώνου. Η Ευρωπαϊκή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να πω συνέβαλε με πολύ χρήσιμο τρόπο στην προσπάθεια με το ψήφισμά του Σαμποτέρο στην ΕΚΟΝ και του Σέρτζιο Κομφεράτη στην ΙΜΚΟ ε, λάμβαμε υπόψη αυτά τα ψηφίσματα. Ε, εργαζόμεθα εντατικά για την αναθεώρηση τη αναλογοδηγία για τις υπηρεσίε πληρωμών. Ένα από τα μέτρα που έχουν προτεραιότητα για την ενία αγορά είναι μια έκθεση για την εφαρμογή του συστήματος πληρωμών. επεσεργαστήκαμε λοιπόν ένα κείμενο, κληρώθηκε με μελέτη αντικτύπου και προβλέπουμε κυρίε και κύριοι, κυρία Πρόεδρε, να εθετέσουμε ένα πακέτο για τι πληρωμέ μέσα Ιουλίου τον επόμενο μήνα με άλλα λόγια που θα περιέχει και την έκθεση εφαρμογής του PST που προβλέπει η οδηγία. Ε, θα συνεχίσουμε λοιπόν με αυτό το συγκεκριμένο θέμα, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με αποφασιστικότητα αλλά χωρίς αυτοσχεδιασμούς και σας ευχαριστώ που με επιτρέψατε να το επαναλάβω αυτό και να το επιβεβαιώσω μπροστά σας σήμερα το πρωί. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε και τώρα το λόγο έχουν οι αγορητές των πολιτικών ομάδων. Υπενθυμίζω ότι δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη διαδικασία της γαλάζιας κάρτας, αλλά δεν προβλέπετε ούτε το ΚΑΣΤΙΑΕ. Για το ΕΛΚ, το λόγο έχει ο κύριος Γκοζές για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε, το Κοινοβούλιο δεν είναι ο αντίπαλος του Συμβουλίου, ούτε είναι ανταγωνιστής είναι συνημοθέτης μαζί με το Συμβούλιο, σε ίσους όρους με το Συμβούλιο. Και υπό αυτή την ιδιότητα παρεμβαίνει σήμερα το Κοινοβούλιο για να διαπιστώσει και να καταγγείλει τις καθυστερήσεις που συσσωρεύονται για την έγκριση απαραίτητων κειμένων. Η Επιτροπή προσπάθησε να προτείνει τα κείμενα για να αντιμετωπιστεί η κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα απευθυνθώ στην Επιτροπή, διότι θεωρώ ότι η Επιτροπή και ειδικότερο ο Επίτροπος Μπαρνιέ έκαναν ό,τι απαιτείτο με τα μέσα που διέθεταν και πρέπει να τον ευχαριστήσουμε γι' αυτό. Βεβαίω, το πρόγραμμα το εκλογικό και ανανέωση επιτροπή καθιστά δύσκολη την έγκριση πριν από το τέλο τη θητείας προτάσεων που θα έρθουν και που είναι πάρα πολύ απαραίτητε. Αυτό που διακυβεύεται εδώ ωστόσο είναι τα κείμενα που έχουν ήδη αποτελέσει αντικείμενο μια συμφωνία στο Κοινοβούλιο και που μπλοκάρονται στο Συμβούλιο. Άκουσα αυτά που είπατε κύριε Υπουργέ. Ε, το Συμβούλιο δουλεύει καλά, ικανοποιητικά, δεν, θέλω να ε, παρουσιάσω έναν κατάλογο των κειμένων που υποφέρουν. Ελπίζω ότι το Συμβούλιο και οι συνεργάτες σας θα βρουν τα απαραίτητα λεπτά για να εξετάσουν το ψήφισμα που θα εγκριθεί την Πέμπτη. Θέλω να επιμείνω στις ε, καταστροφικές συνέπειες ωστόσο της σημερινής κατάστασης. Καταρχήν, μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Το είπα προηγουμένως, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο βρίσκονται πάνω στην ίδια βάση. Χρειάζεται μια ε, ε, ουσιαστική συνεργασία ανάμεσα σε αυτά τα δύο όργανα. Γιατί το Συμβούλιο δεν μπορεί να συμφωνήσει, ενώ στο Κοινοβούλιο, παρόλη την ε, πολιτική του πολυμέρεια και τις διαφορές της εθνικότητές του, βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα, στις διαφορές που μπορεί να προκύψουν. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα που θέτω για την επίλυση της κρίσης που μας μαστίζει παρόλες τις δηλώσεις των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων κάθε φορά που συνεδριάζουν, τα αυτό το μπλοκάρισμα ε, στο Συμβούλιο δείχνει ότι δεν είναι ε, ικανοποιητική η απόδοση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν αν θέλουμε και αν δεν μπορούμε σαν, τις άλλες, σαν χώρες να βγούμε από την κρίση είναι επειδή έχουμε ένα μοντέλο ε, στο οποίο ε, θέλουμε. Γι' αυτό πρέπει να λάβει μέρος της ευθύνη στο Συμβούλιο και να δώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση την ε, αναγκαία όθηση. Αυτό το μπλοκάρισμα δημιουργεί νομική ανασφάλεια και η αναμονή των οι επενδυτές, οι επιχειρηματίες περιμένουν να δουν τι θα συμβεί, τι θα αποφασιστεί, ποιες θα είναι οι αποφάσεις. Δεν μπορούν, μπορούν ωστόσο να, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και να έχουν κείμενα, τα λόμπι που δεν έχουμε εμείς. Πρέπει λοιπόν να δούμε ακριβώς ποια θα είναι η πορεία, η εξέλιξη. Αυτό το μπλοκάρισμα τροφοδοτεί ανεύθυνες αλλά και αποτελεσματικέ δηλώσεις όλων των ευρωσκεπτικιστών κάθε πλευρά, οι οποίοι καταδικάζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, την κατακρίνουν όπως θα το ακούσουμε και άλλες φορές. Αυτό το μπλοκάρισμα δημιουργεί προβλήματα, προβλήματα παραλύει μια επατελεσματική χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Πρέπει λοιπόν να λάβει δράση το Συμβούλιο. Άκουσα μόνο τη μετάφραση, αλλά έχω εμπιστοσύνη στους Γερμινείς. Δεν θα κάνω οποιαδήποτε παρατήρηση για μια αμφιβολία ή περιφρόνησης που διαισθάνθηκα. Ίσως δεν κατάλαβα καλά. Κυρία Πρόεδρε, έφτασε πλέον η στιγμή να προβάλλουμε μια άλλη εικόνα της Ευρώπης και όχι ε, ε, την εικόνα ε, μιας σειράς αυτοκινήτων που διαισθανθηκα ισως δεν καταλαβα καλα κυρια προεδρε εφτασε πλεον η στιγμη να προβάλλουμε μια άλλη εικόνα της Ευρώπης και όχι την, την εικόνα μιας σειρά αυτοκινήτων που εμφανίζονται το βράδυ στο Συμβούλιο για να λάβουν μέρος σε διάφορες συζητήσεις. Είδαμε τι έγινε με την φορολογική απάτη. Δεν μας πιστεύουν, δεν πιστεύουν σε εσά εσά δεν πιστεύουν σε εμά οι ψηφοφόροι, οι πολίτε. Πρέπει λοιπόν να αποκαταστήσουμε τι ζημιέ που προκλήθηκαν από αποφάσει που δεν ανακοινώθηκαν σωστά για την κυπριακή κρίση πρέπει, πρέπει λοιπόν να, να ξεπεράσουμε τα προβλήματα, να αντιμετωπίσουμε ε, αποτελεσματικά την κατάσταση, διότι επέρχονται εκλογές και ε, υπάρχει, υπάρχει, ε, έχουμε το πρόβλημα να προβάλλουμε σε πολύ λίγο διάστημα την εικόνα, τη σωστή εικόνα της Ευρώπης. Είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε και ελπίζουμε ότι θα συμβάλλει και το Συμβούλιο σε αυτή την προσπάθεια. Σας ευχαριστώ οι σοσιαλιστές. Η κυρία Φερέρα έχει το λόγο για δύο λεπτά. Θα μιλήσω αγγλικά, θα μιλήσω θα είναι πιο εύκολο αυτό για το οικονομικό τομέα που ήταν και το επίκεντρο της κρίσης και οι μεταρρυθμίσεις που βρίσκονται υπό εξέλιξη είναι μια προϋπόθεση για την, την αντιμετώπιση και λήξη της κρίσης και να διασφαλίσουμε τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας για την ανάπτυξη. Επανάληψη αυτών των φράσεων. Τώρα όμως πρέπει να γίνει κάτι συγκεκριμένα χειροπιαστά, να δώσουμε αποτελέσματα στους πολίτες. Ξεκίνησε δουλειά και πρέπει να ολοκληρωθεί. Πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί σε αυτά που θα κάνουμε. Ζητούμε από το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Καλωσορίζουμε τα μαντάτα τα οποία μας παρουσίασε ο Επίτροπος Μπαρνιέ για την ολοκλήρωση των εκκρεμουσών προτάσεων για τις ε, τραπεζικές υπηρεσίες και προτάσεις στο δυνατόν γοργότερα ενιαίοι e μηχανισμοί επίλυσης ε, ε, προβλημάτων ε, όσον αφορά τον, το νομοθέτημα για τις ασφάλειες αξιών. Θέλουμε να ολοκληρωθούν αυτά γοργά ώστε να μπορέσουν αυτά τα χαρτοφυλάκια να λάβουν υπόψη και τη θέση του Ευρωκοινοβουλίου. Αναμένουμε λοιπόν διαπραγματεύσεις που πρέπει να ξεκινήσουν με το Συμβούλιο. Κάνουμε λόγο για την εγγύηση των καταθέσεων όμως υπάρχουν αυτά από το Φεβρουάριο του 2012 και κρεμούν το πλαίσιο επίλυση προβλημάτων. Αναμένουμε ακόμα τη δραστηριοποίηση του Συμβουλίου, ακόμα και αν έχει αναγγελθεί ω κύρια προτεραιότητα από το Συμβούλιο αυτό. Περιμένουμε ακόμα μη 2. Αναμένουμε ιδιαίτερα την επιτάχυνση των διαδικασιών για να σημειωθεί πρόοδο προ μια τραπεζική ένωση. Είναι ακρογωνίω λίθος αυτό για το μέλλον. Η υιοθέτηση τη πρότηση για τον ενιαίο μηχανισμό CRD4. Επίση, διαδικασίε όσον αφορά αφορά τις ε, διατάξεις για τις τράπεζες που είναι σημαντικά στοιχεία για την Τραπεζική Ένωση. Για να υπάρξει σταθερότητα και ασφάλεια για τους καταθέτες θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα από ένα ενιαίο μηχανισμό εγγύησης καταθέσεων και ένα ενιαίο πλαίσιο επίλυσης προβλημάτων όσον αφορά τις ε, τράπεζες. Σαφείς κανόνες και κανονισμούς ε, για τη διάσωση τραπεζών θα πρέπει όλα αυτά να καθοριστούν ώστε πλήρως να προστατεύονται όλοι οι καταθέτες σε όλα τα κράτη-μέλη. Και εν τέλει το Ευρωκοινοβούλιο πάντα επομιζόταν τις ευθύνες του για να μπορέσουν να ολοκληρωθούν έγκαιρα και με ευθύνη αυτά τα θέματα. Ο ενίος μηχανισμός ε, εποπτείας. Μέσα σε πολύ στενές προθεσμίες ε, εργαστήκαμε και πρέπει ακόμα να, να αναμένουμε να δραστηριοποιηθεί το Συμβούλιο. Ακόμα αναμένουμε τις διαπραγματεύσεις και την ολοκλήρωση από το Συμβούλιο Μήνυμά μου προ το Συμβούλιο είναι σταματήστε πια τι δηλώσει και τι υποσχέσει. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένε χειροπιαστέ δράσει. Αυτό περιμένουμε. Κυρία Υπουργέ, πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίε και να ολοκληρωθούν τα χαρτοφυλάκια. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ για του πράσινου. Συνάδελφε Γκίγκολτ, έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Συνάδελφοι, κύριε Πίτροπε, πρόεδρε, για να είμαστε σαφέστατοι επ' αυτού του θέματος. Μπορούμε να παριθμίσουμε και πάλι όλα τα χαρτοφυλάκια βέβαια, τα οποία δεν ολοκληρώθηκαν ακόμα από πλευρά του Συμβουλίου και θα το εκτιμούσα αν είχαμε μια άμεση ανταλλαγή απόψεων επ' αυτών. Ο κατάλογος είναι σαφέστατος. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι υπάρχει πρόβλημα το ότι έχει συντάξει προτάσεις γοργά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ένα μεγάλο κατάλογο αναγκαίων προτάσεων και πολλές από αυτές δεν εξετάζονται και δεν ολοκληρώνονται από το Συμβούλιο. Σαφέστατα πρέπει να το πούμε αυτό. Αυτό δεν πιστεύω ότι είναι η ευθύνη της Ιρλανδικής Προεδρίας. Κάνει καλή δουλειά η Ιρλανδική Προεδρία. Γι' αυτό παρακαλώ να μην δημιουργηθεί σύγχυση από αυτές τις επικρίσεις μας. Όμως σε σχέση με το, τις αρνήσεις και αμφισβητήσεις της πραγματικότητας, ποια είναι η πραγματικότητα, δεν καταλήγεται στο να βρείτε στο Συμβούλιο συνένεση και κοινέ θέσεις σε ένα χαρτοφυλάκιο. Τι πρέπει να κάνετε όπως τα βλέπει τα πράγματα το Κοινοβούλιο. Για να μην διαμφισβητηθεί και διακυβευτεί η καλή εικόνα της Ευρώπης, αλλάξτε μέθοδο εργασίας. Θα πρέπει να σταματήσει κανείς να την ευήκονού σε κάποιες προτάσεις κύκλων από τις, τις χώρες από τα κράτη-μέλη. Ξεκινήστε να ψηφίζετε και να ρυθμίζετε τα θέματα όπως το κάνουμε στο Ευρωκοινοβούλιο. Μην αναμένετε και χρονοτριβείτε. Να περάσετε στην ψήφιση προβλημάτων και διευθέτησή τους. Να υιοθετήσετε μια αυθεντικά ευρωπαϊκή μέθοδο. Αυτό αναμένουν οι πολίτες. Δεν είναι αποδεκτό η Λιθουανική Προεδρία η οποία θα ακολουθήσει μετά την Ιρλανδική Προεδρία να ζητεί από το Ευρωκοινοβούλιο να υπάρξουν ιεραρχήσεις αναγκών. Σημαντικά θέματα για τους καταναλωτές ε, όπως τα, τα και πολλά άλλα θέματα θα ακολουθήσουν στην ημερήσια διάταξη νομοθετικά. Πιέζει ο χρόνος. Το πραγματικό θέμα είναι πώς θα αλλάξει την μέθοδο εργασίας του το Συμβούλιο ώστε να μπορέσετε από το Συμβούλιο να καταλήξετε σε συνένεση ή σε μια κοινή θέση τουλάχιστον σε όλα τα θέματα που εκκρεμούν και βρίσκονται στο τραπέζι και περιμένουν οι πολίτες απαντήσεις. Εδώ πρέπει να δραστηριοποιηθείτε. Δώστε μια λύση σε αυτά τα προβλήματα. Μην αρνείστε την πραγματικότητα. Δεχτείτε ότι υπάρχει πρόβλημα και με την Προεδρία και την πείρα σα και την καλή δουλειά που κάνετε μέ στι δομέ που υπάρχουν, να προτείνετε με βάση την πείρα σα μια λύση που μπορεί να υιοθετηθεί σε αυτά τα προβλήματα. Δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι στι χρηματοοικονομικέ υπηρεσίε δεν θα ολοκληρωθεί το χαρτοφυλάκιο σε αυτή τη θητεία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για το ECR. Συνάδελφε Σβίνμπορν, έχετε το λόγο για 1,5 λεπτό. Η χρηματοστική κρίση χρειάζεται και νομοθετική δράση, χρειάζεται και για την εμπιστοσύνη των πελατών επενδυτών, για τη ροή κεφαλαίων εντός και από, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς για την άπτυξη ε, και χρειαζόταν για τι εταιρείε και για τι επενδύσει. Χρειαζόταν εμπιστοσύνη. Όμω, ατελή νομοθεσία δεν μα δίνει ένα μήνυμα εμπιστοσύνη, δημιουργεί αβεβαιότητα και θα αποθαρρύνει τι εταιρείε και τα άτομα και τι μεγάλε εταιρείε από τι αγορέ μα. Προσπαθήσαμε να, από τη διάσκεψη των 20 στο Pittsburgh να ασχοληθούμε με τα παράγωγα ε, μόνο 11 μετέχουμε, ε, επίπεδο 2 δεν έχουμε προχωρήσει καθόλου σε παγκόσμιο επίπεδο και πόρα έχουμε από το να πετύχουμε τι υποχρεώσει, τι εμπορικέ που έχουν θαυτεί σε ένα μύφιτ που έχει πολιτικό χαρακτήρα σε διάφορα χατοφυλάκια στο Συμβούλιο. Αν ξεκινήσουμε την νομοθεσία θα πρέπει να μπορούμε να την ολοκληρώνουμε εγκαίρω. Παράδειγμα, το CSDR, το θέμα του CSDR θα έπρεπε να είναι θετικό μήνυμα, θα έπρεπε να ενθαρρύνει ε, την αγορά να δημιουργήσει αναγκαίες υποδομές και να υπάρχουν και για ε, αναγκαίες υποδομές για το πρόγραμμα που θα ξεκινήσει το 2015. Η ομοφωνία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε από, τη μηχανή, από τον τομέα και τους επενδυτές όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είναι κάτι που θα πρέπει να δημιουργηθεί, αλλά έχουν κολλήσει τα θέματα στο Συμβούλιο. Θα πρέπει να υπάρχουν διαδικασίε για την επίλυση των προβλημάτων και την εξηγήνση όχι μόνο των τραπεζών, αλλά για όλε τι υποδομέ των αγορών, συμπεριλαμβανομένη και, και των διευρυμένων CCP και των CSD βέβαια. Η έλλειψη προόδου όσον αφορά βασικά χαρτοφυλάκια οδηγεί σε έλλειψη εμπιστοσύνη, έλλειψη βεβαιότητα για τι επιχειρήσει σε μια παγκόσμια αγορά και σίγουρα καταλήγει σε έλλειψη εμπιστοσύνη από πλευρά πολιτών μα. Δεν εμπιστεύω τη δυνατότητά μα να μπορούμε να θεσπίζουμε ένα σύστημα που είναι ασφαλέστερο για αυτού. Α κάνουμε λιγότερα αλλά καλύτερα. Σα ευχαριστώ για την ομάδα EFD. Ο κύριος Μπλουμ έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, επίτροπε, ε, κατανοώ κάπως. Πρέπει να πω ότι ε, κατανοώ το Συμβούλιο και, γιατί προσπαθείτε να κάνετε το αδύνατο και το Κοινοβούλιο προσπαθεί να, κάνετε, να πετύχετε το ακατόρθωτο. Όπως γνωρίζουμε στην Αυστρία, για να ρυθμίζει κανείς χρηματοστατικές υπηρεσίες χρειάζεται κανείς τέλεια γνώση της αγοράς και αυτό είναι αδύνατο, δεν μπορεί να γίνει. Ε, καμιά φορά είναι γνωστό ε, σαν η θανατηφόρα αυταπάτη. Θέλουμε να υπάρχει ελευθερία όσον αφορά τη σύναψη συμβάσεων, ούτω ώστε το άτομο, ο επενδυτής, να μπορεί να συνάπτει συμβάσει σύμφωνα των νέων σε μια δημοκρατία που αναγνωρίζει την ιδιοκτησία. Και ο τραπεζίτη, με οποιοδήποτε τραπεζίτη και διαχειριστή επενδύσεων θέλει, χωρί να παρεβαίνει το κράτο και θα πρέπει βέβαια να συνεπάγεται ότι υπάρχει εγγύηση για προστασία των καταναλωτών. Οι τράπεζες κρύβονται πίσω από την νομοθεσία. Και η νομοθεσία τους κρατά εκτός φυλακής όταν εξαπατούν το κοινό. Και εσείς τελικά στην όλη συνωμοσία συμμετέχετε. Βγει, να βγείτε από την περιοριστική νομοθεσία για όνομα του Θεού και αφήστε τον τόπιο νόμο να ακολουθήσει το δρόμο του. Ευχαριστώ πολύ. Για την ΚΟΕ, ο κύριος Κλούτο έχει το λόγο για ένα λεπτό. Μάλιστα, ευχαριστώ. Συνάδελφοι, επιτόπου με πολίτες και εκλογής όταν μιλάει κανείς, ρωτάνε κατά το πέμπτο έτος της κρίσης τι είναι αυτό που κάναμε εμείς ως πολιτικοί να αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση. Στο πέμπτο έτος αυτής της κρίσης για να αντιμετωπιστεί επιτέλους μπορούμε να πούμε ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεκάδες χαρτοφυλάκια νομοθετικά έχουμε ολοκληρώσει. Πιστεύω ότι στο Ευρωκοινοβούλιο, ακόμα και όταν έχουμε διαφορετικέ απόψει σε κάποια θέματα, σε πολλέ περιπτώσει καταλήγουμε σε λογικέ ε, προτάσει προ όφελο των πολιτών. Αυτό κάνουμε τουλάχιστον. Εκπονούμε λογικέ προτάσει προ όφελο των πολιτών. Δεν κατανοούν όμω οι πολίτε γιατί όλα αυτά δεν περνάνε σε εσά και λέμε Εντάξει, τα περισσότερα από αυτά τα οποία εκπονούνται στο Κοινοβούλιο τροχοπεδούνται στο Συμβούλιο. Και αυτό δεν το καταλαβαίνουν οι πολίτε. Γιατί τροχοπεδούνται στο Συμβούλιο. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο κατεπηγόντω πρέπει να επιλύσουμε. σω αυτή η καθυστέρηση την οποία έχουμε μπροστά μα και για την οποία συζητάμε σήμερα το πρωί έχει κάποια σχέση με την αδιαφάνεια των εργασιών στο Συμβούλιο. Με μεγαλύτερη διαφάνεια στι εργασίε του Συμβουλίου, ίσω οι λόγοι για αυτέ τι καθυστερήσει θα ήταν πιο διαφανεί. Θα αποκαλυπτόντουσαν και αυτό τουλάχιστον θα βοηθούσε κάπω του πολίτε να κατανοήσουν το τι συμβαίνει στο Συμβούλιο. Θα άνοιγε έτσι μια δυνατότητα να καταλάβουν τα αίτια αυτών των καθυστερήσεων και να καταπολεμηθούν αυτά τα αίτια των καθυστερήσεων. Ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε γοργή και καλή θετική λύση του προβλήματο. Και υπό το δικό μα πρίσμα καλό θα ήταν αν τα χαρτοφυλάκια που εκκρεμούν μέχρι το τέλο τη θητεία, τη κοινοβουλευτική μας θητείας θα μπορούσαν να ολοκληρωθούν. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Το λόγο έχει Επίτροπος, ο κ. Μπαρνιέ. Κυρία Πρόεδρε, κύριε και κύριοι, κυρίες και κύριοι βουλευτές, δεν θα ξαναρχίσω ολόκληρη τη συζήτηση, αλλά σε αυτό το σημείο θέλω να επιβεβαιώσω δύο πράγματα. Τη διαθεσιμότητα, τη δική μου, του επιτελείου μου, της γενικής μου διεύθυνσης, των συνεργατών μου, δουλεύουμε με μια μικρή ομάδα αλλά ιδιαίτερα αποτελεσματική για να διευκολύνουμε πέρα από την υποβολή προτάσεων να προτείνουμε στρατηγικές και να διευκολύνουμε επίσης το έργο του Συμβουλίου Υπουργών, στο οποίο συμμετέχω τακτικά, το έργο του Κοινοβουλίου, σεβόμενος την αυτονομία και την κυριαρχία σας και συμμετέχοντας επίσης με χρήσιμο τρόπο στους τριμερείς διαλόγους που είναι τόσο πολύ σημαντικοί. Ε, αναφέρω αυτή τη διαθεσιμότητα ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτό που είχαμε αναγγείλει. Είναι θέμα αποτελεσματικότητας για την οικονομική σταθερότητα, για να θέσουμε πιο υγιείς και διαφανείς βάσεις και πέρα από τη διαφάνεια και την υπευθυνότητα να υπάρξει και λίγη ηθική και δεοντολογία που είχαν χαθεί για να θέσουμε στην υπηρεσία της πραγματικής οικονομίας τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και όχι το αντίθετο όπως συνέβαινε για πάρα πολύ καιρό, αυτό κάνουμε και είναι και θέμα αξιοπιστίας για το G20, για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, για μας ως ευρωπαϊκοί θεσμοί να δείξουμε ότι μπορούμε, ότι μπορούμε να εφαρμόσουμε, να υλοποιήσουμε αυτά που λέμε στην, για να προωθήσουμε την οικονομία στην Ήπειρό μας. Ε, ε, ε, όπως και ο, Σουίν, ο κύριος Σουίνμπορ, έχουμε αντιμετωπίζουμε σε οικονομικό επίπεδο μια τεράστια παγκόσμια κρίση. Βεβαίω, έχουμε... Η κρίση προήλθε, υπήρχε το θέμα του χρέους στην Ευρώπη, αλλά η κρίση μας ήρθε από την, ε, τις Ηνωμένε Πολιτείες και το G20 το G20 ήταν εκείνο που δημιούργησε αυτό το πρόγραμμα το οποίο να ακολουθούμε. Πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε ότι οι μεγάλοι εταίροι του G20 που είναι καταρχήν οι Ηνωμένε Πολιτείε, 80% των συναλλαγών είναι υπερατλαντικές συναλλαγές. Πρέπει λοιπόν παράλληλα ο καθένα με τους νόμους μας να εφαρμόζουμε το ίδιο πρόγραμμα. Κυρίε και κύριοι, αφιερώνω πάρα πολύ χρόνο για 8 φορά εδώ και τρία χρόνια θα πάω στι Ηνωμένε Πολιτείε να εξασφαλίσω ότι υπάρχει αυτό το level playing field, ίσοι κανόνε για όλου, σε συνεργασία με του σημαντικότερου εταίρου. Σα ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Το λόγο έχει η Υπουργό η κυρία Κράιτον. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Βασική προτεραιότητα τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω είναι να προωθήσει βιώσιμη οικονομική ανάκαμψη, δημιουργήσει της απασχόλησης Και νομίζω ότι αυτός είναι κοινό μας στόχος Και για να πετύχουμε τον ελόγο στόχο, θα πρέπει να έχουμε δραστηριοποίηση ενεργό και συνεργασία μεταξύ όλων των θεσμικών οργάνων, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και άμεσα πρέπει να έχουμε συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Καλή νομοθεσία αποτελεί κοινή προσπάθεια όλων των τριών θεσμικών οργάνων και πολύ συχνά είναι θέμα ευαισθητών ε, συμφωνιών που πρέπει να πετύχουμε και πρέπει να το καταλάβετε. Πέρασα 5,5 μήνες παίζοντα το ρόλο της Προέδρου στην Προεδρία και είναι πάρα πολύ οδυνηρό, πάρα πολύ δύσκολο να πετύχει κανεί την ευαίσθητη συνένεση ε, και εντό των θεσμικών οργάνων και μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Ομαλή και επικοδομητική συνεργασία είναι το κλειδί, ούτω ώστε να πετύχουμε τα ευκταία αποτελέσματα και αυτή είναι η κοινή μα πρόκληση. Ε, καταρτίζοντας προτεραιότητες μας, προσπαθήσαμε να εξισορροπήσουμε την αναγκαιότητα να ανταποκριθούμε σε κατα... κατεπίγουσες νέες ανάγκες που διαφάνησαν ε, λόγω της κρίσης και από την άλλη να το εξισορροπήσουμε με την θέμα αντιμετώπισης διαθωτικών θεμάτων όπου οι νομοθέτες προσπαθούν να δουν πέρα από το άμεσο μέλλον και θέλουν να πετύχουμε βιώσιμη ανάκαμψη και υψηλά ε, επίπεδα απασχόλησης, να μειωθεί η υψηλή ανεργία. Ε, συνεργαστήκαμε με το Κοινοβούλιο, στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πετύχαμε αποτελέσμα σημαντικό τομέα όπως είναι οι χρηματοστητικές υπηρεσίες και θα συνεχίσουμε άοκνες προσπάθειες σε αυτά τα χαρτοφυλάκια. Ήδη συνεργαζόμαστε βεβαίως με τους συναδέλφους της επικείμενης Λιθουανικής Προεδρίας και εσείς γνωρίζω ότι το κάνετε αυτό και θα εξασφαλίσουμε μια συνέχεια της προσέγγισης που ακολουθεί το Συμβούλιο στα διάφορα χαρτοφυλάκια που θεωρούμε σημαντικότατα. Ξέρω ότι συνάδελφος στην ελληνική κυβέρνηση, ο, ο Υπουργός Μάικλ θα είναι συνεδρία της Επιτροπής ΕΚΟΝ στις 24 ε, Ιουνίου για μια αξιολόγηση του τέλους της Προεδρίας και μια αναθεώρηση που θα είναι μια καλή ευκαιρία να αναθεωρήσουμε τη σημαντική πρόοδο που επετεύχθη όσον αφορά αυτά τα ζητήματα, κάτι που περιέγραψα λεπτομερέστερα στα εισαγωγικά μου σχόλια. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω, μέλη του Κοινοβουλίου, ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προωθήσουμε το πρόγραμμα των χρηματοστατικών υπηρεσιών στο δεύτερο εξάμεινο του 2013 και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εξασφαλίσουμε το ότι θα διατηρηθεί η όλη ορμή των προσπαθειών που νομίζω ότι είναι κάτι που πετύχαμε τους τελευταίους μήνες και το περιέγραψα στα εισαγωγικά μου σχόλια. Αυτό που θα ήθελα να πω κλείνοντας είναι ότι ευχαριστώ την Sharon Bowles και την Επιτροπή Οικονομικών και Σμουτικών Θεμάτων. Ήταν έξοχη συνεργασία μας, νομίζω ότι πετύχαμε πολλά. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Μισελ Μπαρνιέ και την ομάδα του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έξοχη συνεργασία. Δεν ήταν εύκολα, είχαμε τα προβλήματά μα. Νομίζω ότι πετύχαμε ουσιαστική πρόοδο. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μα, σίγουρα. Πολλά μέλη το ανέφεραν αυτό. Και νομίζω ότι όλοι μας τα διάφορα θεσμικά μας όργανα πρέπει να διπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας και να εργαστούμε επικοδομητικά και ε, συνεργάσιμα τους επόμενους μήνες ούτως ώστε να πετύχουμε όλους τους κοινού μας στόχους και κυρίως πριν από τις ευρωεκλογές του επόμενου έτους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Λάβαμε μία πρόταση ψηφίσματος ε, στο τέλος της συζητήσεως, περατώθηκε η συζήτηση και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο στις 12. Τώρα θα έχουμε κάποια λεπτά διάλειμμα στον αφορά τη εργασία μα πριν ξεκινήσει η συζήτηση για το επικείμενο συμβούλιο.